ο θα έρθει ο κύριο Αβραμόπουλο στην έδρα. Πρέπει να εξετάσουμε την έκθεση Χαλάχο για το Ευρωπαϊκό Ταξιδιωτικό Έγγραφο για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκών τρίτων χωρών. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή για πέντε λεπτά. Euh, Ευχαριστώ. Όπως γνωρίζουμε η Ευρώπη δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχής στα θέματα της κρίσης των μεταναστών και των προσφύγων. Ένα τμήμα της εξήγησης της αποτυχίας είναι η έλλειψη πολιτικής επιστροφής. Η ανικανότητά μας να στείλουμε πίσω αυτούς των οποίων απερίφθηκε η αίτηση να μείνουν στην Ένωση. Μόνο το 40% ε, των αποφάσεων αυτών επιστροφής τελικά σε κάποια φάση εφαρμόζονται. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπονομεύει την αξιοπιστία του συστήματος χορήγησης ασύλου. Είναι κάτι το οποίο ενθαρρύνει επίσης και την κατάχρηση του συγκεκριμένου συστήματος από αυτούς οι οποίοι δεν ε, χρειάζονται διεθνή προστασία και ε, στην ουσία ξοδεύουμε και δεν έχουμε πόρους για να καλύψουμε τις ανάγκες αυτών που έχουν ανάγκη από την διεθνή αυτή προστασία. Υπάρχουν λοιπόν εδώ κάποια συγκεκριμένες προτάσεις για την επιστροφή των συγκεκριμένων αυτών ανθρώπων. Οι ρυθμίσεις οι οποίες ισχύουν βέβαια σήμερα δεν γίνονται δεκτές από τις χώρες στις οποίες προορίζονται οι άνθρωποι αυτοί και δεν πληρούνται επίσης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συμφωνιών που θα έπρεπε να ισχύουν. Υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις σε σχέση με τη φύση της πρότασης αυτής και στο Κοινοβούλιο και εκτό Κοινοβουλίου. Με ρώτησαν πολλοί αν δεν θα είναι δυνατό να ζητήσει κανείς προστασία στην Ένωση και αν όλοι οι μετανάστες θα απελαθούν. Όχι βέβαια. Μιλάμε για μια τεχνική πρόταση η οποία δεν αφορά τους κανόνες τους σχετικούς με το άσυλο, με την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή με την έκδοση των συγκεκριμένων ταξιδιωτικών εγγράφων. Το θέμα είναι η εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας. Ο κανονισμός αυτός είναι ένα μικρό κομμάτι, σημαντικό όμως θα έλεγα, του συστήματος ασύλου, διότι μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μας ε, στον τομέα των επιστροφών. Ε, θα μειώσει επίσης ε, το διοικητικό και γραφειοκρατικό άχθος και για τις χώρες μέλη της Ένωσης και για τις χώρες τελικής, τελικού προορισμού ε, έχουν τεθεί ορισμένα θέματα στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου. Σαν παράδειγμα εμείς ε, διατηρήσαμε ε, την δυνατότητα η αναγνώριση των ταξιδιωτικών εγγράφων να είναι τμήμα των διαπραγματεύσεων με τις χώρες επανεισδοχής. Το Κοινοβούλιο επίσης κράτησε τη συγκεκριμένη αναφορά του άρθρου 19 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για τα παιδιά και την ανάγκη τήρησης των διεθνών υποχρεώσεών μας. Η συμφωνία αντικατοπτρίζει επίσης και τις παρούσες ισχύουσες απόψεις για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Το ταξιδιωτικό έγγραφο αυτό δεν είναι μία μαγική λύση δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό η έλλειψη ενός εναρμονισμένου εγγράφου είναι η πραγματική αιτία πίσω από την άρνηση των χωρών επανεισδοχής. Ένα σημαντικό στοιχείο της συμφωνίας είναι να διασφαλίσουμε την πλήρη αναθεώρηση ε, του εγγράφου αυτού ε, πέρα από την προβλεπόμενη ε, περίοδο δύο χρόνια μετά από τη θέση σε ισχύ οπότε ε, τότε θα ενταχθεί στην κανονική οδηγία. Η συμφωνία υπογραμμίζει την ανάγκη να αναζητήσουμε το έγγραφο επιστροφής στα πλαίσια των συμφωνιών που θα υπογράψει η Ένωση και οι χώρες μέλη με τρίτες χώρες. Για να πετύχουμε τον στόχο αυτό είναι απαραίτητο το νέο έγγραφο να χρησιμοποιηθεί πλήρως από όλες τις χώρες μέλη. Μέσω της ενημέρωσης των μέσων τα οποία έχουμε βαδίζουμε ε, προς μια κατάσταση που θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, διασφαλίζοντας ένα ποσοστό επιστροφών αποτελεσματικό. Αυτή η συμφωνία είναι ένα καλό αποτέλεσμα για το Κοινοβούλιο και σε σχέση με το μέλλον. Ένα έγγραφο το οποίο θα χρησιμοποιείται ευρύτερα από τα κράτη-μέλη και θα αναγνωρίζεται ευρύτερα και από τρίτες χώρες. Θα ήθελα να ολοκληρώσω ευχαριστώντας την Προεδρία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους τους χειώδεις εισηγητές για τη συνεργασία και τις προτάσεις τους και το αποτελεσματικό έργο σε αυτό το νομοθετικό χαρτοφυλάκιο. χαρτοφυλάκιο. Ελπίζω, ευελπιστώ ότι θα μπορέσετε να υποστηρίξετε ψηφίζοντας, υπερψηφίζοντας αυτήν την πρόταση. Θα λάβει τώρα τον λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Πράγματι, τώρα θα λάβει τον λόγο ο κύριος Επίτροπος, ο κύριος Αβραμόπουλος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική επιστροφή των παρανόμως διαμενών των μεταναστών είναι είναι το επιστέγασμα μιας ε, αποτελεσματικής και επιτυχούς πολιτικής για τη μετανάστευση. Είναι εξίσου θεμελιώδες για την διατήρηση της εμπιστοσύνης από τους πολίτες μας για το πώς χειριζόμαστε τα θέματα μετανάστευσης και επίσης ε, αντιμετωπίζει τα θέματα της ε, μη ασφαλούς και παράτυπης μετανάστευσης. Το θέμα του, των ταξιδιωτικών εγγράφων ήταν ένα από τα κύρια προσκόμματα που παρεμπόδιζαν την ε, αποτελεσματική επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί με ένα έγγραφο ταξιδιωτικό που θα υποκαθιστά το κανονικό ταξιδιωτικό έγγραφο και που θα εκδίδεται από τα κράτη-μέλη. Για να είναι έγκυρο όμως και να χρησιμοποιείται όπως πρέπει, αυτό το έγγραφο πρέπει να αναγνωρίζεται από τρίτες χώρες. Υπήρξε ένα πρότυπο για ένα τέτοιο ε, πρότυπο ταξιδιωτικού εγγράφου για τις απελάσεις ε, ε, υπηκόων παρανόμως διαμενόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1994. Όμως τα κράτη-μέλη δεν κάνουν χρήση συχνά αυτής της δυνατότητας. Οι χώρες εκείνες με τις οποίες υπάρχει η διαπραγμάτευση για συμφωνία επανεισδοχής ασκούν επικρίσεις ότι δεν είναι ικανοποιητικές οι πτυχές ασφάλειας και υπάρχει η δυνατότητα πλαστογράφησης ε, και παραχάραξης αυτού του εγγράφου. Γι' αυτό πρότεινε μια, ένα κανονισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ρυθμιστούν αυτά τα θέματα, θεσπίζοντας ένα νέο ταξιδιωτικό ευρωπαϊκό έγγραφο για την επιστροφή ε, υπηκών τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα δημιουργήσει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πρότυπο με διευρυμένε ε, τεχνικές δυνατότητες όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας. Ιδιαίτερα θα συμμορφώνεται με επακριβή, επακριβή στοιχεία που αφορούν την ασφάλεια ελαχιστοποιώντας κινδύνους παραχάραξης και πλαστογράφησης και για να μην δημιουργηθούν επιπρόσθετα προσκόμματα και επιβάρυνση γραφειοκρατική τα χαρακτηριστικά ασφάλειας θα ακολουθούν εκείνα τα χαρακτηριστικά που ήδη υφίστανται σήμερα στα ε- ταξιδιωτικά έγγραφα που αφορούν επίσης και θεωρήσεις. Θα υπάρχει ένα ασφαλές πλαίσιο για αυτό το έγγραφο που θα διευκολύνει την αποδοχή αυτού του ε, ταξιδιωτικού εγγράφου από τις τρίτες χώρες. Αυτό είναι ένα σημαντικό τεχνικού χαρακτήρα μέσο το οποίο θα βοηθήσει ώστε να ενδυναμωθεί αυτό η δυνατότητα αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έπρεπε να θεωρείται ως ένα στοιχείο μεταξύ πολλών άλλων που πρέπει να προαχθούν. Αποτελεί μέρος, τμήμα μιας ευρύτερης στρατηγικής που δημιουργείται με το πρόγραμμα δράσης για τις επιστροφές και εδώ υποστηρίζονται και οι προσπάθειες των κρατών μελών για την επιστροφή και επανεισδοχή των παρανόμως διαμενών των υπηκών τρίτων χωρών με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, ιδιαίτερα και τον σεβασμό των διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον εισηγητή μας, τον κύριο Χαλαχαχό, και επίσης τις ευχαριστίες μου προς τους σκιώδεις εισηγητές της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστώ. Ξεκινάνε τώρα οι πολιτικές ομάδες. Κύριε κυρία Μουσολίνη, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το να εγγυηθούμε την, ε, τον επαναπατρισμό με ταχύ τρόπο, με διαφανή τρόπο των παράνομα μεταναστευόντων είναι προϋπόθεση ούτω ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και υποδοχή και να δώσουμε προστασία στους νόμιμους μετανάστες. Ακριβώς γι' αυτό, σε αυτό το πολύ κανονισμό δεν μπαίνει τίποτα καινούριο, αλλά απλώς επικαιροποιούμε το έγγραφο του 1994. Το είπε και ο εισηγητής. Τον ευχαριστώ για τη δουλειά του. Διευκολύνεται η αναβάθμιση των προτύπων, αποφεύγουμε τις ε, πλαστογραφήσεις και μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι τα τρίτα κράτη να αναγνωρίσουν το έγγραφο αυτό, το ταξιδιωτικό αυτό έγγραφο. Να σταματήσω, να σταθώ μια στιγμή ε, σε κάτι που απασχόλησε το ΕΛΚΑ, κυρίως την ομάδα του ΕΛΚΑ, και που αφορά το άρθρο 24 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για τους ανήλικους. Είναι ένα θέμα το οποίο φυσικά με απασχολεί πάρα πολύ. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω λοιπόν ότι εμεί κάνουμε συγκεκριμένη αναφορά στο γεγονός ότι σε όλε τι πράξει που αφορούν τους ανήλικους τα έγγραφα που τους δίνουν οι δημόσιοι θεσμοί και οι ιδιωτικοί φορείς θα πρέπει πάνω απ' όλα να προστατεύουμε τα συμφέροντα του ανήλικου. Επομένως, ακόμα και αν αυτό είναι ένας κανονισμός τεχνικός, θελήσαμε να βάλουμε στον κανονισμό αυτό αυτό το σημαντικό απόσπασμα. Νομίζω λοιπόν ότι έγινε μια θαυμάσια δουλειά, ε, συνεισέφεραν όλοι και εμείς είμαστε υπέρ της έγκρισης του κανονισμού αυτού και επαναλαμβάνω ότι είναι αυτό ένα πρώτο βήμα προς μια καλύτερη δυνατότητα υποδοχής των, νομίμως, ε, των νόμιμων μεταναστών και με μια πιο ταχεία διαδικασία απέλασης των παρανόμων διαμενόντων. Κυρία Νταλή, για δύο λεπτά τους σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ. Οι πολιτικές ε, για την μετανάστευση πρέπει να συναποτελούνται από διάφορες συνιστώσεις, ε, ακόμα και την μετεγκατάσταση και την ε, ε, μεταφορά των μεταναστών. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας και πρέπει να επιστρέψουν στην χώρα προέλευσής τους. Φυσικά πάντα αντιμετωπιζόμενοι με αξιοπρέπεια και με σεβασμό των δικαιωμάτων τους. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για μας τους δημοκράτες. Έτσι το σύστημα επιστροφής ε, σε σχέση με τους ε, ε, μετανάστες και η αναγνώριση του εγγράφου, του ταξιδιωτικού εγγράφου που δεν είναι ευρύτερα αποδεκτό από αρχές τρίτων χωρών για διάφορους λόγους και δημιουργούνται προβλήματα μεγαλύτερο πλαίσιο διασφάλισης ε, και των εγγράφων και των μηχανισμών επιστροφής των παρανόμων διαμενόντων, παρανόμως διαμενόντων μεταναστών θα διευκολύνει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών ώστε να, μπορούν να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων ε, κατά τις διαδικασίες επιστροφής και επανεισδοχής αυτών των μεταναστών. Με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων ιδιαίτερα και των ανθρωπιστικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των παιδιών. Τώρα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή όλων αυτών και σε σχέση και με το ταξιδιωτικό έγγραφο για την επιστροφή των μεταναστών αυτών με εφαρμογή και των διμερών ακόμα ε, συμφωνιών. Δεν θα επιλύσει αυτό το ταξιδιωτικό έγγραφο ε, τα προβλήματα μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι όμως ε, ένα λιθαράκι ένα, μια συνεισφορά για να αντιμετωπιστεί η ευρύτερη κρίση μετανάστευση. Θέλω να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο για τη συνεργασία του. Ένα λεπτό κύριο Στίβεν από το ECR. Η κυρία Στίβεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Πράγματι πρέπει να ρυθμιστεί η ιστορία αυτών οι οποίοι ε, πρέπει να εγκαταλείψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποσοστό επιστροφής όμως δεν ξεπερνά το 30% νομίζω. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μια αποτελεσματική πολιτική επιστροφής είναι απαραίτητη. Οι μετανάστες από τρίτες χώρες και ιδιαίτερα από αφρικανικές χώρες θα πρέπει να σταλούν πίσω στις χώρες τους. Κάτι τέτοιο όμως ε, δυσκολεύεται από το ότι δεν έχουν ε, έγγραφα ταξιδιωτικά. Παίρνουν κάποια προσωρινά έγγραφα τα οποία πλαστογραφούνται όμως πάρα πολύ εύκολα και οι χώρες προορισμού αρνούνται να δεχτούν την εγκυρότητά τους. Και γι' αυτό λοιπόν ο κανονισμός αυτός έχει σημασία γιατί προτείνει πράγματι ένα ενιαίο έγγραφο το οποίο θα είναι ε, δύσκολο να πλαστογραφηθεί και θα βοηθήσει μια αποτελεσματική πολιτική επιστροφής. Η έκδοση των εγγράφων αυτών θα πρέπει να ανήκει στα κράτη-μέλη φυσικά. Πεσέρα Μπαστερέτσεα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Κύριε Επίτροπε, όταν κάνουμε λόγο για την επιστροφή υπηκών τρίτων χωρών που παραμένουν παράνομα παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνουμε λόγο για το ταξιδιτικό έγγραφο για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της ασφάλειας στις επιστροφές. Όμως εδώ έχουμε έλλειψη συντονισμού και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εκείνοι οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για διεθνή προστασία πρέπει να επιστρέψουν. Όμως θα ήθελα να συμμεριστώ την ανησυχία για εκείνους που άδικα ε, επιστρέφουν επειδή αποτυγχάνει η κοινή πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση. Ξέρουμε το τι συμβαίνει σε σχέση με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν στις χώρες τους ε, αυτά τα άτομα και τι γίνεται σε σχέση με τη διεθνή προστασία. Και κάθε λεπτό που περνάει επιδεινώνεται η κατάσταση. Παραβιάζονται αυτές οι αρχές και από την Τουρκία σε σχέση και με τα παιδιά και τις έγκυες γυναίκες. Και όταν ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες ε, που, στις οποίες ε, υπάρχει άμεση απειλή του Ισλαμικού κράτους και πείτε μου κύριε Επίτροπε θεωρούμε πραγματικά μια ασφαλή χώρα την Τουρκία για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες ή σε σχέση με τα σύνορα της Ισπανίας είχαμε δεκάδες Σαχαριανούς που με βίαιο τρόπο επεστράφησαν στο Μαρό Μαρόκο στο φράχτη στα σειρματοπλέγματα της Μελίγια. Και αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί κυρίες και κύριοι. Είναι πραγματικά ε, επιτακτική ανάγκη να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Αντιμετωπίζει όμως μια κατάσταση παράλυσης η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθύνουμε έκκληση ε, ώστε να μπορέσει να γίνει κάτι εν ώψη της απραξίας ε, του Συμβουλίου των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή ενωμένη Ευρώπη. Αλλά χρειάζονται χρειάζονται τη βοήθειά μας οι πιο ευάλωτοι ε, πολίτες, εκείνοι που διαφεύγουν, προσπαθούν να φύγουν από τη βαρβαρότητα και τη δυστυχία. Ευχαριστώ. Περίμενα να ακούσω το τέλος της ε, διερμηνίας. Μιλούσατε πάρα πολύ γρήγορα. Ήθελα να διορθώσω ότι μιλάτε εξ ονόματος των φιλελεύθερων. Διορθώ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χθε κάναμε μια συζήτηση για την επόμενη συνοδοκορυφή του ΟΗΕ για τη μετανάστευση. Η κυρία Μογκερίνη ζήτησε από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να, αναλάβουν τι ευθύνε του απέναντι σε αυτού που χρειάζονται διεθνή προστασία. Με αυτό το υποτιθέμενο ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο δεν θα προχωρήσουμε. Στην πραγματικότητα θέλουμε να παρακάψουμε ε, τα προβλήματα που ε, αντιμετωπίζουμε από τρίτες χώρες οι οποίες αρνούνται να δεχτούν αυτά τα άτομα. Όταν ακούμε τις ε, μαρτυρίε των μεταναστών που είναι όλο και περισσότερο ε, θύματα αστυνομική βίας, διερωτώμε για το σεβασμό των, θέληση ε, της των ατόμων που απελάφνονται. Το ελάχιστο θα ήταν τα έγγραφα αυτά να συντάσσονται σε γλώσσα που καταλαβαίνουν. Γι' αυτό υποβάλαμε μια τροπολογία και ελπίζω να την περάσετε, γιατί δεν είναι ελάχιστο αυτό. Επίσης, οποιαδήποτε συμφωνία με τρίτη χώρα η οποία ε, δέχεται πολύ περισσότερους πρόσφυγες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλό θα ήταν να, να τη δούμε, να δούμε τι κάνει η τρίτη αυτή χώρα πριν ε, κλείσουμε εμείς ε, το ελεφάντινο πύργο μας. 1,5 λεπτό, ο επόμενος ομιλητής. Κύριε Σαρτζεντίνη, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Μία πολιτική επιστροφή είναι φυσικά απαραίτητη για να συμπληρωθεί η πολιτική ασύλου. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ε, πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες τους έχουν ανάγκη από ταξιδιωτικά έγγραφα, σύγχρονα ταξιδιωτικά έγγραφα με φωτογραφία αποφεύγοντας την δυνατότητα πλαστογράφησης. Η πράσινη είναι κατά όμως γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αναλύσει τις επιπτώσεις αυτής της πρότασης απλά προβλέπει ενίσχυση της πολιτικής επιστροφής. Το θέμα είναι να πείσουμε τις τρίτες χώρες να υποδεχθούν εκ νέου τους πολίτες τους. Κάτι το οποίο δεν είναι μόνο απαραίτητο για ένας, γιατί ένας μεγάλος αριθμός αυτών των ανθρώπων δεν θέλουν να επιστρέψουν, αλλά και γιατί οι περισσότερες από τις χώρες αυτές δεν θέλουν να τους υποδεχθούν. Συνεπώς λοιπόν έχουμε να κάνουμε με χώρες οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα δημοκρατικές και πολλές φορές θα χρησιμοποιήσουν και με παράλογο τρόπο, με μη νόμιμο τρόπο, τα ιδιωτικά δεδομένα που θα έχουν στη διάθεσή τους μέσω του νέου συστήματος. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνονται όλο και πιο κατασταλτικές. Ήδη από το καλοκαίρι του 2015 ακολουθούμε τον λάθος δρόμο. Άρνοτ 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όταν βλέπετε τον τίτλο της συζήτησης αυτής, όταν κάποιος βλέπει τον τίτλο της ε, συζήτησης αυτής, θα μπορούσε να πιστέψει ότι πρόκειται για ανθρώπους που ήρθαν ε, νόμιμα στην Ένωση, αλλά παράνομα συγγνώμη στην Ένωση, έτσι και αλλιώς δεν θα μπορούν να σταθούν πλέον και να παραμείνουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά βέβαια οι στόχοι πολλές φορές ε, έχουν σαν μοναδική θα έλεγα μοναδικό χαρακτηριστικό την έννοια της εναρμόνισης και γι' αυτό οι προτάσεις αυτές είναι διακοσμητικές και δεν αλλάζουν πραγματικά τις αποφάσεις οι οποίες εφαρμόζονται τώρα και οδηγούν σε περισσότερη παράνομη μετανάστευση. Εμείς θα τηρήσουμε στάση αποχής γιατί η απόφαση αυτή πρώτον δεν θα ισχύσει για το Ηνωμένο Βασίλειο έτσι κι αλλιώς. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αυτό που θα αποφασίσει τι νόμους θα εφαρμόσει και θα ήταν υποκριτικό για μένα να θέλω να παίρνω μέρος σε τέτοιες αποφάσεις που δεν θα φορούν στη χώρα μου σε λίγο καιρό. Το θα απόσχω από αυτή την ψηφοφορία. Φοντάνα, 2,5 λεπτά από το EFDD. Ευχαριστώ. Είμαστε ενώπιον ενός ψηφίσματος που θα μπορούσαμε να το δούμε και θετικά. Δηλαδή, μετά από πολλά χρόνια, βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θεωρεί ότι τα άτομα τα οποία φτάνουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που, εν πάση περιπτώσει, δεν πλήρουν τα κριτήρια ούτω ώστε παραμείνουν στο εσωτερικό τη Ένωση, θα πρέπει να επαναπατριστούν. Το πρόβλημα όμω είναι ότι δεν θα ήθελα, όπω τόσε άλλε φορέ συνέβη, να μείνουμε στα ευχολόγια, να κάνουμε κάποια πράγματα, όμω τελικά φτιάχνουμε απλώ γραφειοκρατία που θα δυσκολεύσει ακόμη περισσότερο τα Υπουργεία των κρατών μελών. Επίτροπε, πέρυσι ξεκινήσαμε, κάναμε μια απόπειρα να βάλουμε μια τάξη στη μετανάστευση. Μην ξεχνάτε ότι μέχρι τώρα, το 2016, φτάσαν στην Ιταλία πάνω από 100.000 άτομα. Το ξέρετε σίγουρα. Το 60% από τα άτομα αυτά ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν έχουν κανένα κριτήριο για να δικαιούνται να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειάζονται τι διεθνού προστασίε. Δεν φεύγουν από πολέμου. Δεν δικαιούνται λοιπόν την προστασία αυτή και παρόλα αυτά επαναπατρίστηκαν λιγότερο από 5.000 άτομα. Μόνο 5.000 άτομα επαναπατρίστηκαν ε, πραγματικά. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν. Ε, υπάρχει και πολιτικό επίσης πρόβλημα, πρόβλημα πολιτικής βούλησης. Αν κάποιος πιστεύει ότι πρέπει να δεχτούμε τους πάντες, αλλά ξέρουμε ότι τόσα εκατομμύρια ανέργων ε, που έχουμε στην Ευρώπη, πώς θα δώσουμε, πώς θα εξασφαλίσουμε μέλλον στους ανθρώπους αυτούς. Επομένως αυτά τα άτομα δεν μπορούν να ενταχθούν στις κοινωνίες μας. Και αυτό τι συμβαίνει όταν δεν εντάσσονται συμβαίνει, σημαίνει ότι μερικοί θα πάνε σε εγκληματικέ δραστηριότητε, ορισμένοι θα τρελαθούν ας πούμε, θα, μπουν στον, ε, θα πάνε στην Ισλαμική τρομοκρατία, τα έχουμε δει αυτά. Επομένως, για την ε, επιβίωση της Ευρώπης χρειάζεται μια σοβαρή πολιτική επαναπατρισμού. Ελπίζω να υπάρχει και η πολιτική βούληση να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί υπάρχουν τόσε αντιδράσει και θα εκφραστούν αυτέ. Γιατί ιδεολογικά, α πούμε, υπάρχουν διάφορα άτομα τα οποία θεωρούν ότι πρέπει να έρθει όλο ο κόσμο στην Ευρώπη. Όλοι η Αφρική. Οι πάντε στην Ευρώπη. Ξέρετε όμω αυτό είναι ιδεολόγημα. Δεν γίνεται. Και δυστυχώ τα ιδεολογήματα μα καταστρέφουν. Ελπίζω πραγματικά λοιπόν να μείνει αυτή η πρόθεση. Ελπίζω να βρεθεί μια λύση, αλλά προσοχή, προσοχή. Θα πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά γρήγορα και με αποτελεσματικέ μεθόδου. Γιατί Εάν δεν το κάνουμε έτσι το πράγμα, ο κίνδυνος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, για, ακριβώς για το λόγο της μετανάστευση, θα εκραγεί. Κύριε Φωντάνα, μιλούσατε, ε, εκφράζετε το ΙΕΝΕΦ. Γκάμπριελ. Έλκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Επίτροπο. Συνάδελφοι, σήμερα έχουμε να κάνουμε με ένα συγκεκριμένο μέσο, ένα τεχνικό μέσο, το οποίο όμως μπορεί να βοηθήσει να συμπληρωθούν κενά στην πολιτική ασύλου. Γι' αυτό και θα στηρίξω την συγκεκριμένη πρόταση. Ε, θα ήθελα να τονίσω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις δράσεις μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναδιαπραγματευτούμε, αναδιαπραγματευτούμε συμφωνίες επανεισδοχής με τρίτες χώρες και γι' αυτό ακριβώς είναι προϋπόθεση να υπάρχει το ε, έγγραφο αυτό σαν ε, ε, τμήμα της διαπραγμάτευσης. Θα πρέπει επίσης να ζητήσω από τα ευρωπαϊκά όργανα να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να συναυθούν συμφωνίες με τον Ήγυρα και την Ιγυρία και ίσως και κάποιες άλλες χώρες στην υποσαχαρική Αφρική είναι περισσότερο απαραίτητο. Θα πρέπει επίσης να ενταχθεί ένα έγγραφο ένα αντίγραφο του εγγράφου αυτού στο Eurodac και στο SIS και θα ήθελα η Βουλγαρία να έχει πλήρη πρόσβαση στο SIS. Έχουμε εξωτερικά σύνορα με την Τουρκία και θα πρέπει να εκπληρώσουμε όλα τα τεχνικά κριτήρια. Πώς θα το πετύχουμε αυτό. Τέλος να υπογραμμίσω ότι το άρθρο 13 της Συμφωνίας του Κοτονού προβλέπει ότι οι χώρες εταίροι μας θα πρέπει να δέχονται τους πολίτες τους, να υποδέχονται πίσω τους πολίτες τους. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το ενιαίο ταξιδιωτικό έγγραφο είναι κάτι το θετικό. Από την άλλη βέβαια δεν μπορεί να καλύψει πλήρως τις απαιτήσει που υπάρχουν έτσι ώστε και οι τρίτες χώρες να εκδίδουν τέτοιου είδους ταξιδιωτικά έγγραφα. Γι' αυτό λοιπόν απαιτείται συνεργασία και με τις προξενικές υπηρεσίες. Πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα μετανάστευσης που αντιμετωπίζουμε. Είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αρκεί να βελτιώσουμε τις τεχνικές παραμέτρους, αλλά αυτό το συγκεκριμένο είναι ένα καλό βήμα. Βάιντεν δύο λεπτά, Πρόεδρε, Επίτροπε. Η Ευρώπη λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφύγων που αντιμετωπίζει. Είναι σημαντικό να δώσουμε βοήθεια για αυτούς τους ανθρώπους σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και μέσα στη θετική καλή παράδοση της έκφρασης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό χρειάζονται σαφείς κανόνες, αποτελεσματικές δομές και τακτές διαδικασίες Απουσιάζουν όμως πολλαπλά αυτά στην Ευρώπη. Κυρίως στα κράτη-μέλη η κατάσταση είναι συγκεχημένη και δημιουργεί ανασφάλεια και αβεβαιότητα για πολλούς ανθρώπους χρειάζεται μια σωστή επισκόπηση και διαφάνεια. Πρέπει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η Ευρώπη και θα πρέπει διοικητικέ διατάξεις και ρυθμίσεις να ληφθούν γι' αυτό. Κυρίως να γνωρίζουν οι άνθρωποι τι θα συμβεί με αυτούς και τι πρόκειται να γίνει. Τα έγγραφα, ταξιδιωτικά έγγραφα για τους παράνομους ε, μετανάστες είναι ένα σημαντικό στοιχείο μέσα στο πλαίσιο αυτό. Ένα τέτοιο ταξιδιωτικό έγγραφο είναι αναγκαίο ώστε η ευρωπαϊκή διαδικασία χορήγησης ασύλου να είναι αξιόπιστη. Πρέπει να είναι ανοιχτή η χρήση αυτού του εγγράφου σε όλους εκείνους που την χάνουν αρνητικής ε, απόφασης όσον αφορά την αίτηση χορήγησης ασύλου. Οι απελάσεις λοιπόν πρέπει να είναι πάντα σύμφωνες με τις αρχές ε, της ανθρωπιστικής και του διεθνούς δικαίου. Χρειάζονται σαφείς νομικές βάσεις. Αυτή εδώ η ρύθμιση είναι ένα τέτοιο στοιχείο. Όταν αυτό το Ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο για την επιστροφή θα προβλέπει διαδικασίες ασφαλής και προδιαγραφές ασφαλής όσον αφορά και την προσυπογραφή συμφωνιών και την έγκριση κρατών. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια Κέρμερ, ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και εγώ υποστηρίζω ρητά την έκθεση του συναδέρφου μας Ράχο και θεωρώ ότι είναι αποφασιστική σημασίας λιθαράκι σε ένα συνολικό μοσαϊκό για να έχουμε μια αποτελεσματική πολιτική ασύλου. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι <clears throat> δεν έχουμε την δυνατότητα απεριόριστα να δεχόμαστε ανθρώπους στην Ευρώπη. Για να υπάρχει χώρος για εκείνους που πραγματικά χρειάζονται αυτή την ε, ε, διαδικασία ε, εγκατάστασής τους και προστασίας τους στην Ευρώπη πρέπει εκείνοι που είναι παράνομοι να επιστραφούν. Γι' αυτό χρειάζεται το ταξιδιωτικό αυτό έγγραφο. Γι' αυτό πρέπει το δυνατόν ταχύτερα να εφαρμοστούν αυτές οι προτάσεις. Και χαίρομαι για το ότι για το θέμα της μετανάστευσης ε, και της πολιτικής ασύλου προχωρούμε στην Ευρώπη προπαρασκευάζοντας ένα τέτοιο σημαντικό μέτρο το οποίο πρέπει όμως να εφαρμοστεί. Δηλαδή χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια συνοδευτική διαδικασία και μια αξιολόγηση για το τι θα γίνεται στα κράτη-μέλη στη συνέχεια. Είναι πολύ σημαντικό όχι στη θεωρία να δράσουμε αλλά πρακτικά χειροπιαστά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τα ευρωπαϊκά κράτη είναι θύματα μιας μεταναστευτικής ροής ενός κύματος χωρίς προηγούμενο. Πρέπει όμως να υπερασπιστούν την ταυτότητά τους. Άργησε να το καταλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και η κυρία Μέρκελ και αντέδρασε λάθος ανοίγοντας τις θύρες. Τώρα όμως φυσικά επανέρχονται σε αυτήν την απόφαση. Διαφωνώ όμως με το ταξιδιωτικό έγγραφο που προτείνεται ναι μεν θα μας επιτρέψει να επαναπροωθήσουμε τους μετανάστες εκτός Ευρώπης, θα είναι ένα διαβατήριο προσέκδοση μόνο που θα ισχύει μόνο για ένα ταξίδι, το ταξίδι της εξόδου. Αλλά από την άλλη θα είναι ένα έγγραφο υπερεθνικό, εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αξιόπιστη. Θα συνεχίσει να υποκύπτει στα λόμπι της μετανάστευσης εμείς θα καταπολεμήσουμε την μετανάστευση όταν ξαναβρούμε την πλήρη μας εθνική κυριαρχία. Ευχαριστώ κύριος Διαστεμέρα, 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, είναι μια καλή νομοθετική πρωτοβουλία αυτή. Συγχαίρω επίσης και τον φίλο Γιούση Άχο ως εισηγητή ε, αυτόν τον κανονισμό. Κανονισμό που εισάγει βελτιώσεις όπως αυτές που ακολουθούν. Εναρμονισμό μέτρων ασφάλειας. Ε, περιορισμό της περίοδου αναμονής ε, παλινόστησης. Συντονισμό ώστε να υπάρχει ένα σύστημα παλινόστησης επιστροφής με περισσότερα χέγγια, με περισσότερα, περισσότερες Ιδιαίτερα προστατεύοντας εκείνους που πρέπει να, να τύχουν τέτοια προστασία επίσης σε σχέση με τις προξενικές αρχές και επίσης ε, θα δυσχεραίνει την πλαστογράφηση και παραχάραξη του εγγράφου αυτού. Όμως οι παράνομοι ε, μετανάστες βλέπουμε ότι πολλές φορές αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης από τις μαφίες και αυτό πρέπει να το ε, παρεμποδίσουμε. Χρειάζεται μια πολιτική στεναρή των, της επανεισδοχής και της επιστροφής και αυτό απαιτεί και μια στεναρή πολιτική για το άσυλο. Ε, ε, μία ένα από τα τροτά σημεία που έχει ο κανονισμός είναι η δυσκολία για την ε, αναγνώριση από τρίτες χώρες. Εδώ είναι κάτι το οποίο εκκρεμεί αυτή η υπόθεση. Πιστεύω όμως Πρόεδρε ότι θα είναι ένα χρήσιμο στοιχείο ώστε ο μηχανισμός για, την τον οποίο είμαι εισηγητής να μπορέσει να προαχθεί. Ευχαριστώ. Κύριε Ντίας Ντεμέρα, υπάρχει ένα ερώτημα, μια μπλε κάρτα, τη δέχεστε. Τον κύριο Φουντσούλη. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ντίας Ντεμέρα, αντιμετωπίζουμε μια, αυτή την κατάσταση τέτοια που το ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο δεν αναγνωρίζεται από τις περισσότερες χώρες που πρέπει να δεχθούν πίσω τους υπηκόους τους. Πώς λοιπόν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Σε πολλές ευκαιρίες αρνούνται να δεχτούν το άτομο αυτό γιατί λένε ότι λείπουν κάποια έγγραφα ή δεν αναγνωρίζουν διάφορα έγγραφα όπως και το ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατάσταση, αυτό το πρόβλημα. Παρακαλώ, ο κύριος Δίας Δεμέρα. Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας, κύριε Φρονζουλίτσα, μια ερώτηση πάρα πολύ σκόπιμη. Τι θα κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις να ενεργοποιηθεί η διπλωματική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει και πρέπει να δραστηριοποιήσει το δυναμικό της στο διπλωματικό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε οι συμφωνίες σε σχέση με τρίτες χώρες ε, να μπορέσουν να προαχθούν για την αναγνώριση αυτού του ταξιδιωτικού εγγράφου. Ελπίζω να απάντησα στο ερώτημά σας. Ο κύριος Λόπεθ Αγιλάρ, 1,5 λεπτό παρακαλώ. Χουάν Φερνάντεθ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το 2014 τα κράτη-μέλη εξέδωσαν 500.000 τέτοιες εντολές επιστροφής από τις οποίες περίπου 200.000, ένα 40% εκτελέστηκαν είναι σε σχέση με τη ρητορική λάθος όταν λένε κάποιοι ότι εισέρχεται οποιοδήποτε και οι επιστροφές δεν λειτουργούν. Όχι, λειτουργούν. Τώρα, η απουσία ενός ε, ενιαίου εγγράφου και ισχυρού αποδεκτού εγγράφου που θα διασφαλίζει ενιαίες διαδικασίες όσον αφορά την ταυτοποίηση των ατόμων που επιστρέφουν είναι μια δυσκολία για να γίνονται δεκτά αυτά από τρίτες χώρες. Το δεχόμαστε αυτό ως προϋπόθεση και η πρωτοβουλία της Επιτροπής είναι θετική. Πρώτα απ' όλα αυτή η πρωτοβουλία να διασφαλίζει πλήρως τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων που καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων άσχετα από την προσωπικότητα, άσχετα από το άτομο. Δεύτερον, να διασφαλίζεται ότι δεν θα γίνονται επιστροφές ατόμων όπου υπάρχει ομοία αντιμετώπιση, όπου υπάρχουν βασανιστήρια και άλλα προβλήματα γιατί δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τέτοιου είδους επιστροφές. Ιδίως θα πρέπει να αλλάξει η αρνητική προσέγγιση από πλευράς της Ευρώπης σε σχέση με τις επιστροφές. Δεν μπορεί να είναι η πανάκια η επιστροφή αλλά ένα μέτρο ίστα της ανάγκης και ίστα της χρήσης για να μην παραμένουν στην Ευρώπη εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να παραμένουν σε αυτήν. Όμως το να αλλάξει η πολιτική για τη μετανάστευση είναι κάτι επιτακτικά αναγκαίο Ευχαριστώ. Κύριος Μπάρεκοφ, ένα Σας ευχαριστώ πολύ προς τον κύριο εισηγητή. Θα ήθελα να πω ότι όσο το δυνατόν νωρίτερα η Ευρώπη μπορέσει να απελευθερωθεί από τους ε, παράνομους μετανάστες, τόσο ταχύτερα θα προχωρήσουμε. Στη Σόφια, 100 μέτρα από την προεδρική κατοικία, υπάρχει μια συνοικία που την αποκαλούν μικρή Βαγδάτη. Στη Βουλγαρία αυτό, στη Σόφια έχει μετατραπεί σε ένα αυτοκινητόδρομο, σε ένα διάβλο παράνομων μεταναστών η Βουλγαρία που περνάνε από την Τουρκία στη χώρα αυτή. Η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να υπερασπιστεί τους πολίτες μας και υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ Μέρκελ και Ερντογάν που δημιουργεί αυτή την κατάσταση και αυτά τα προβλήματα. Πρέπει να δεχθούμε ε, ότι είναι δικοί μας πολίτες ε, οι νόμιμοι μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα μας. Οι παράνομοι πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες τους. Πρέπει να υπερασπιστούμε την Ευρώπη, ιδιαίτερα τα σύνορα μεταξύ της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Πρέτσελ παρακαλώ, δύο λεπτά. Κυρίες και κύριοι, πρόεδρε, κύριε επίτροπε, για πρώτη φορά, έτσι φαίνεται εδώ, περνάμε με πλειοψηφία προς την κατεύθυνση επιστροφών παράνομα διαμενόντων στην Ευρώπη υπηκών τρίτων χωρών που κατέβαλαν προσπάθεια να έρθουν στην Ευρώπη και να τύχουν ασύλου. Αυτό είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα βέβαια. Όμως αφεαυτού δεν επιλύει τίποτα αυτόματα θα πρέπει οι τεχνικές προδιαγραφές να δημιουργηθούν και για ένα ευρωπαϊκό έγγραφο ε, ταξιδιωτικό αλλά και άλλες προϋποθέσεις που πρέπει να υλοποιηθούν. Καταρχήν πρέπει να ασκηθεί πίεση στις χώρες, τρίτες χώρες, ώστε να αποδεχθούν αυτό το έγγραφο να το αποδέχονται. Γιατί χωρίς πίεση αμφιβάλλω αν θα δεχτούν ένα τέτοιο ταξιδιωτικό έγγραφο αυτές οι χώρες. Μπορεί κανείς για παράδειγμα την άσκηση, την πίεσης ε, να την συνδέσουμε με την χορήγηση αναπτυξιακής βοήθειας προς αυτές τις χώρες ή και διαμορφώνοντας αντίστοιχα τις εμπορικές μας σχέσεις ως Ευρώπη με τις χώρες αυτές. Δεύτερον, και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό, πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση στις ευρωπαϊκές χώρες που θα προσθεθεί ως στοιχείο για να επιτευχθεί αυτή η διαδικασία απελάσεων και μπορώ να πω ότι στη Γερμανία η πολιτική βούληση απουσιάζει. Εκεί όπου θα μπορούσαν να γίνουν απελάσεις πολύ συχνά δεν γίνονται. Και για τον συνάδελφο των Σοσιαλδημοκρατών, όπως ανέφερε πιο πριν, η επιστροφή ότι είναι το ίστατο μέσο, το ακραίο ίστατο μέσο, εδώ διαφωνώ κάθετα μαζί του. Δεν είναι ο στόχος του ασύλου να επιτρέπει την μετανάστευση. Η επιστροφή είναι ο ανώτατος στόχος για οποιονδήποτε που εισέρχεται στην Ευρώπη για να τύχει ασύλου, όταν δεν υπάρχει λόγος χορήγησης ασύλου, η για άσυλο, τότε είναι υποχρέωσή μας να επιστρέφονται αυτοί στις χώρες τους και να εντάσσονται σε αυτές. Ο κύριος Βόμποντα, 1,5 λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υποστηρίζω αυτό το, αυτή την απόφαση για το κοινό ταξιδιωτικό έγγραφο για τους υπηκόους τρίτων χωρών που βρίσκονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό είναι να μπορούμε να βελτιώσουμε τα εργαλεία μας για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τους παράνομα διαμένοντες. Γιατί χωρίς ε, λειτουργικά εργαλεία και τα υπόλοιπα στοιχεία της πολιτικής ε, μετανάστευσης δεν θα λειτουργούν επίσης. Στον τομέα της μετανάστευσης και της πολιτικής για τη μετανάστευση οι λύσεις δεν είναι απλές. Αυτό το έγγραφο φυσικά από μόνο του δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα μιας αποτελεσματικής πολιτικής επιστροφών, αλλά θα βελτιώσει την κατάσταση. Καθώς και οι συμφωνίες ε, επανεισδοχής και αυτές ε, θα βοηθήσουν στο βαθμό που συνάπτονται και που υπάρχει να δούνε και λαβήν με αυτές τις τρίτες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν για να, να αναγκάζουμε τις τρίτες χώρες να αναγνωρίζουν αυτό το έγγραφο. Και α στάσουμε τώρα στην εξωτερική πολιτική. Δεν υπάρχουν εύκολε και μεμονωμένε λύσει. Μια αποτελεσματική πολιτική επιστροφών δεν σημαίνει ότι μειώνονται τα πρότυπα της σύμβασης της Γενέβης που οπωσδήποτε πρέπει να τη σεβαστούμε. Και αυτό το τονίζω. Καθώς και να σας πω ότι υποστηρίζω αυτή την προσπάθειά σας. Ο κύριος Μάμικινς για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάθε χώρα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκδιώξει αυτούς οι οποίοι έχουν μπει παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μέτρο το οποίο προτείνεται όμως δεν είναι πάρα πολύ κατανοητό. Αυτοί οι οποίοι δεν είναι πραγματικοί πρόσφυγες γνωρίζουν ότι χωρίς διαβατήριο μπορεί να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για δεκαετίες τέτοιου είδους εμπειρίες φυσικά γίνονται προσπάθειες και από τους υπόλοιπους να αποκτηθούν. Οι πόροι οι οποίοι απαιτούνται για να βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί, ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι φεύγουν, προσπαθούν να ξεφύγουν από τα βασανιστήρια και τους πολέμους, είναι πολύ περιορισμένοι. και δυστυχώς υπάρχει και πολιτική εκμετάλλευση του φαινομένου αυτού πολλές φορές και από τους ίδιους τους πολιτικούς. Δεν αρκεί λοιπόν το να εκδώσουμε ε, κάποια ταξιδιωτικά έγγραφα. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή και ο κανονισμός αυτός μπορεί ίσως να βοηθήσει να βελτιωθεί το σύστημα. Δεν είναι όμως πανάκια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε με αυτόν τον κανονισμό για αυτό το ταξιδιωτικό έγγραφο η πολιτική επιστροφών είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος ε, για την πολιτική μετανάστευση. Είναι όμως ένα, ένας ευάλωτος κρίκος ε, και σε σχέση ε, e για την εντολή να εγκαταλείψουν οι παράνομοι. Όμως 40% επιστρέφουν από αυτούς στη χώρα προέλευσης τους ή στη χώρα από την, από την οποία πέρασαν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει εδώ να δούμε ότι εφόσον δεν επιτρέπεται να βρίσκονται εδώ 60% δηλαδή πάνω από το ίμιση δεν επιστρέφουν και έτσι δεν τους αφορούν οι κανόνες και η νομοθεσία μας μπορούν να παραμένουν λοιπόν από ό,τι φαίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το δοκούν. Θα πρέπει λοιπόν να οδηγούμαστε σε ένα μικρότερο ποσοστό ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η πολιτική επιστροφών και να είναι η όλη δράση μας για τις ε, παλινοστήσεις και τις, ε, την επανεισδοχή τους και τις επιστροφές να παράσχουμε και ένα πλαίσιο υποστήριξης ε, και οικονομικά να δράσουμε ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει το σχέδιό μας για αυτές τις επιστροφές. Εκείνοι οι οποίοι ζητούν προστασία και αξίζουν αυτής της προστασίας πρέπει να μπορούν να μείνουν στην Ευρώπη. Λιμπεράς και ένα λεπτό. Επίτροπε, καλωσορίζω αυτή την πρωτοβουλία. Έχω μία ερώτηση. Γιατί δεν το κάναμε αυτό νωρίτερα. Νομίζω αν το είχαμε κάνει πριν από ένα χρόνο θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Πολλά προβλήματα τα οποία μας πνίγουν τώρα δεν θα υπήρχαν καν. Πρέπει να διαφοροποιήσουμε ανάμεσα αυτούς που μένουν εδώ παράνομα αλλά που η ζωή τους κινδυνεύει από, νόμιμα συγγνώμη, αλλά που ζωή τους, και που ζωή τους κινδυνεύει από τους παράνομους μετανάστες. Πολλοί δεν έχουν έγγραφα γιατί τα έχουν πετάξει. Το γεγονός ότι δεν έχουν έγγραφα δεν σημαίνει ότι, έχουν, ότι είναι στο απειρόβλητο και ότι μπορούν να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώ το αντίθετο θα πρέπει να συμβαίνει. Θα πρέπει, αν έχει έγγραφα, να διευκολύνεται η παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα ο κύριος Γιούνκερ έκανε την ομιλία του την ίδια μέρα με αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα. Την ομιλία για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μ' αρέσει αυτό, αυτή η πρωτοβουλία και θα υπερψηφίσω αυτή την πρωτοβουλία. Ο κύριος Σόγκορ, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βελτιώσουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά ασφάλειας των ατόμων που διαμένουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των εγγράφων δηλαδή, των ατόμων αυτών. Πιστεύω ότι τα άτομα σε παράνομη κατάσταση δεν θα μειωθεί, ο αριθμός δεν θα μειωθεί με τη βελτίωση αυτού του εγγράφου. Νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε δύσκολα προβλήματα. Τι θα κάνουν οι αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν ένας ετών άσυλο, όπου του έχουμε αρνηθεί το, το άσυλο, δεν θέλει να επιστρέψει και βάζοντα σε κίνδυνο μερικέ φορέ και τη ζωή του για να αποφύγει την, ε, τον επαναπατρισμό του. Τι θα κάνουμε με αυτά τα άτομα. Αυτά τα άτομα προσπαθούν να αποφύγουν πάση θυσία την απέλαση. Αυτό δεν είναι και να μας καταπλήσει. Θα κάνουν τα πάντα οι άνθρωποι αυτοί για να παραμείνουν στην Ευρώπη. Το ερώτημα λοιπόν που σας ε, υποβάλλω είναι πώς είναι δυνατόν να εφαρμόσουμε την απόφαση άρνησης του ασύλου. Εάν όλοι παραμείνουν, όλοι όσοι διαφεύγουν από τον κίνδυνο και όσοι δεν έχουν κανένα λόγο να παραμείνουν εδώ, παραμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι πολιτική μετανάστευση αυτή, είναι χάος. Χάος. Επίσης, οι τρίτες χώρες ε, μερικές φορές δείχνουν προθυμία για να δεχτούν τους πολίτε πολίτες αυτούς τους τρίτων χωρών. Γιατί δεν έχουν ε, δεδομένα, γιατί δεν υπάρχουν ταξιδιωτικά έγγραφα κτλ. Μερικές φορές τις κατανοούμε. Νομίζω όμως και ότι η εκτέλεση των αποφάσεων απέλασης θα δυσκολέψουν και τις αρχές των κρατών μελών. Πρέπει να αποφασίσουμε τάχιστα. Πάμε στο Catch the Eye. Κινίτσι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το φαινόμενο το μεταναστευτικό έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Απαιτείται μια νέα πολιτική η οποία να περιλαμβάνει και την δυνατότητα καλύτερης ρύθμισης μέσω ενός νομοθετικά αναγνωρισμένου εγγράφου το θέμα του επαναπατρισμού αυτών που παραμένουν παράνομα στην Ευρώπη. Μια τέτοια αποτελεσματική πολιτική θα μας επιτρέψει να φροντίσουμε καλύτερα αυτούς που χρήζουν διεθνούς προστασίας, ιδιαίτερα τις πιο εύθραυτες κατηγορίες όπως τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Αυτό θα αυξήσει το επίπεδο ασφάλειας, θα μειώσει τη γραφειοκρατία ε, και νομίζω ότι για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η Επιτροπή πρέπει να ξεκινήσει ένα επικοδομητικό διάλογο με τις τρίτες χώρες σε επίπεδο επανεισδοχής. Είναι απαραίτητο θα έλεγα οι διαδικασίες αυτές να γίνονται με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φυσικά να καλύψουμε όλα τα δικαιώματα των ανηλίκων. Ο κύριος Συναδεινός, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση θα είχε ιδιαίτερη σημασία αν η Ένωση διέθετε τη βούληση και την αποφασιστικότητα να δώσει λύση στο πρόβλημα της λαθρομετανάστευση. Εξηγώ. Είναι αδύνατο να παραβλέψουμε ότι στο έδαφος της Ένωσης υπάρχουν εκατομμύρια παράνομα διαμένοντε μετανάστες και άτομα των οποίων η αίτηση για χορήγηση ασύλου έχει απορριφθεί. Όλοι αυτοί διαμένουν ή κυκλοφορούν παράνομα. Είναι ανόητο να πιστεύουμε ότι το μεγάλο πρόβλημα για την επαναπροώθησή του είναι η χορήγηση σωστών ταξιδιωτικών εγγράφων στην κοροϊδία της τουρκίας και των υπολείπων τρίτων χωρών που έχουν υπογράψει συμφωνίες επανειστοχής δεν τις τηρούν και μάλιστα απαιτούν περισσότερα ανταλλάγματα οφείλουμε να απαντήσουμε δυναμικά. Αφενός χρειάζεται αποτελεσματική φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης από τα κράτη μέλη όπου θα εισέρχονται μόνο όσοι τηρούν τα διεθνή πρότυπα και αφετέρου διακοπή κάθε επαφή συζήτηση και συνδιαλλαγή με όποια τρίτη χώρα δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα. τέλο για όσους συνεχίζουν λογοπαίγνια με τη χρήση του όρου παράτυπη μετανάστευση έχω να δηλώσω το εξής είναι παράλογο στο ίδιο κείμενο να χρησιμοποιείς τον όρο παράνομα διαμένοντες αλλά παράτυπα εισελθόντες μετανάστες. ευχαριστώ. nezakonita migracija jedan je od gorućih problema s kojim se hitno moramo pozabaviti. toleriranje nezakonite migracije i prihvaćanje da je na neki način neizbježna Ένα από τα πιο καυτά θέματα είναι και πρέπει εδώ να δώσουμε προσοχή στο ότι ε, ανεχόμαστε τους παράνομους. Πολύ σκληρά εργαζόμενοι άνθρωποι θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη και να μπορέσουν να ζήσουν σε αυτήν και δεν μπορούν να το καταφέρουν διότι υπάρχει τεράστια γραφειοκρατική επιβάρυνση. Όμως εξακολουθούμε να αφήνουμε ανθρώπους που δεν έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα να παραμένουν στην Ευρώπη. Το νέο αυτό ταξιδιωτικό έγγραφο σε σχέση με την επιστροφή επιστροφή όλων αυτών είναι ένα σωστό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση. Θα μειώσει την γραφειοκρατική επιβάρυνση σε σχέση με τα κράτη-μέλη και θα παράσχει και εγγυήσει. Ωστόσο όμως εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα δώσει τα ευκταία, τα επιθυμητά αποτελέσματα αν δεν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το πρόβλημα των παρανόμων μετανάστων. Grazie, signore Presidente ο απαράδεκτα μεγάλος αριθμός παρανόμων μεταναστών που κατακλείζουν όλες τις χώρες της Ευρώπης και κυρίως της Ελλάδος ή συναλληφθούν άμεσα μέτρα προκειμένου αυτοί να απελαθούν. Υπό την έννοια αυτή η τροποποίηση του υφισταμένου ταξιδιωτικού εγγράφου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα ως μια απλή τυπική διαδικασία. Εάν οι παράνομοι μετανάστες κατορθώσουν να βρουν τρόπους για να παραμένουν στις χώρες της Ευρώπης, τότε θα προσελκύσουν και άλλους ομοίους τους να έρθουν εδώ. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μεταξύ αυτών που έρχονται παράνομα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης υπάρχουν επικίνδυνοι τζιχαντιστές και σκληροί τρομοκράτες οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τόσα ιδεχθή εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει. Πρέπει με πάση θυσία να προστατεύσουμε την ασφάλεια των λαών των χωρών της Ευρώπης και να αδιαφορήσουμε για λόγους σκοπιμότητος στις πιέσεις των διεθνών κυκλωμάτων εκμεταλλεύσεως μεταναστών καθώς επίσης και στις ε, ε, γραφικές αντιδράσεις των απανταχού αλληλεγγύων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έχει ζητήσει το λόγο και ο κύριος Μαριάς αλλά δεν είναι εδώ. Γι' αυτό θα περάσουμε στην απάντηση του κύριου Επιτρόπου. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές. Επιτρέψτε μου να αρχίσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου για αυτή την πολύ γόνιμη συζήτηση και τι παρατηρήσει που ακούστηκαν. Όπω είπα και στην αρχή των εισαγωγικών μου παρατηρήσεων, αυτό το ταξιδιωτικό έγγραφο είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τις ε, πολιτικές επιστροφών και για να γίνουν αυτές πιο αποτελεσματικές. Όμως δεν είναι το μόνο μέσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εργαστεί τώρα για την υλοποίηση των διαδικασιών σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη για να επιτευχθεί ο στόχος. Ο στόχος είναι να προαχθεί η επανεισδοχή ή και άλλες συμφωνίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών με ευρύτερη αποδοχή αυτού του ταξιδιωτικού εγγράφου από τρίτες χώρες. Αν στοχοθετήσουμε, τις, ε, στοχεύσουμε τις ενέργειές μας σωστά θα μπορεί να είναι ένα εργαλείο με σημαντική ε, εμβέλεια για, την, ε, για τις χώρες για την επιστροφή των προσφύγων αυτών. Όπως ζητήθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναφέρεται στο Συμβούλιο και θα αναφέρεται και στο Κοινοβούλιο για την εξέλιξη αυτών των διαδικασιών ε, σε δύο, μετά από δύο χρόνια. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να τονίσω ότι δεσμευόμεθα εμείς να υποστηρίξουμε τη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή ο Γενικός Διευθυντής μας βρίσκεται στη Βουλγαρία, στη Σόφια, για διαπραγματεύσεις, διαβουλεύσεις με τις βουλγαρικές αρχές και για να αξιολογηθούν οι ανάγκες των Βουλγάρων. Και όσον αφορά και τη χρηματοδότηση και συνοριοφύλακες και όλα τα άλλα θέματα, όπως τόνισε και ο πρόεδρος Γιούνκερ σήμερα στον λόγο για την κατάσταση της Ένωσης που εξεφώνησε. Αυτή η έκθεση θα είναι άμεσα διαθέσιμη. Είναι προτεραιότητα αυτή η πρωτοβουλία για και για μένα προσωπικά. Σας ευχαριστώ και πάλι για την υποστήριξή σας Ευρωβουλευτές, για την εξαιρετική συνεργασία για αυτό το νομοθετικό ζήτημα. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής, ο κύριος Χάλα Αχώ. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις συνεισφορές σας. Θα ήθελα σύντομα να απαντήσω σε κάποια από τα πιο κρίσιμα σχόλια και της αριστεράς και της δεξιάς. Υπάρχουν τεράστιες ιδεολογικέ διαφορές για το τι πρέπει να κάνουμε με την παράνομη μετανάστευση και με τη μεταναστευτική πίεση. Πιστεύω παρόλα αυτά ότι περισσότερο συμφωνούμε ότι η ισχύουσα νομοθεσία θα πρέπει να εφαρμοστεί. Αυτός ο κανονισμός αφορά ακριβώς αυτό. Έχουμε κανόνες σε ό,τι αφορά τον άσυλο και την παραμονή. Αν ένα άτομο μπορεί de facto να παραμείνει ανεξάρτητα από το αν ε, συντρέχουν οι προϋποθέσεις, τότε δεν υπάρχει λόγος να έχουμε κανόνες. Όπως είπα, αυτό είναι επιζήμιο και για την αξιοπιστία της νομοθεσίας μας και ενθαρρύνει όλο και περισσότερους ανθρώπους να περάσουν τη Μεσόγειο. Παρότι και εγώ είμαι ευρωσκεπτικιστής και δεν υποστηρίζω μια, ένα συγκεντρωτικό σύστημα ε, διεκπαιρέωση των αιτήσεων ασύλου. Παρ' όλα αυτά, συμφωνώ με αυτό το έγγραφο γιατί είναι συμβασμό. Πιστεύω ότι το ταξιδιωτικό έγγραφο είναι παράδειγμα συνεργασία που δίνει προσθέμενη αξία στι προσπάθειε των κρατών μελών, ανεξάρτητα από τι πολιτικέ αποφάσει που παίρνουν σε εθνικό επίπεδο. Σα ευχαριστώ λοιπόν πολύ, συνάδελφοι, επίτροπε και βασίζομαι στην υποστήριξή σα αύριο. Ευχαριστώ. Πέρα στη συζήτηση.